με σειρματόσχηνα. Να ακούσουμε πρώτα την συγγήτρια κυρία Φόρντ. Θα αναφερθώ στα μέσα ατομικής ε, προστασίας. Ε, πραγματικά έγινε μια ενδιαφέρουσα μελέτη εν σχέση με την ε, εσωτερική αγορά και πώς ε, διαμορφώνεται στις 28 χώρες μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έπρεπε να αντιδράσουν. Είναι πριν από μερικές εβδομάδες πολλοί από εμά είδαν ε, σοκαριστικές εικόνες μιας, ενός εργοστασίου στην ε, Τουρκία που παράγει ψεύτικα ε, σωσίβια σωσίβια μαϊμούδες και τα οποία όποιος τα φορά έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να πνιγεί. Άρα λοιπόν προκειμένου να εμποδίσουμε επικίνδυνα προϊόντα να μπουν στην ευρωπαϊκή αγορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διατύπωσε κοινέ ε, προδιαγραφέ που καλύπτουν ε, κάσκες, σωσίβια, το είδο ατομικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε διάφορους χώρους εργασίας επίσης. Επίσης όταν χρειάστηκε να ε, προστατευθεί, ε, ένα συλλεκτικό ε, προσωπικό από την μετάδοση ιών. Ε, και τέτοιου είδους προδιαγραφές ε, διευκολύνουν τις αρχές να ανοιχνεύσουν τα επικίνδυνα προϊόντα και να τα απομακρύνουν από την αγορά. Οι κοινέ προδιαγραφές στην Ευρώπη μπορεί επίσης να βοηθήσουν τους ε, κατασκευαστές στις πωλήσει του σε άλλα μέρη του κόσμου. Οι τεχνικές μεταβολές, στην, οι τεχνικές αλλαγές στην έκθεση που συζητούμε σήμερα θα προσθέσουν και θα εξυγχρονίσουν 25 έτη προηγούμενες νομοθεσίες και αυτό θα βοηθήσει τους ε, κατασκευαστές ε, καθώς και τους προμηθευτές και τους καταναλωτές. Ωστόσο, ένα από τα βασικά στοιχεία της κοινή αγοράς ε, είναι το επίπεδο των προδιαγραφών. Πόσο ψηλά θα πρέπει να ε, τοποθετηθεί ο γνώμονας. Θεωρώ ότι ένας, ε, μια νέα νομοθεσία θα πρέπει να βασίσει μια ξεκάθαρη ανάλυση κόστους ε, ωφέλειας και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει επαρκής μελέτη αντικτύπου. Δεν πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το τι φοράμε σπίτι μας για παράδειγμα για να πλύνουμε τα πιάτα οι πολιτικοί θα πρέπει να βγουν από την ε, κουζίνα, όχι να εκπονούν πολιτικές εν σχέση με το πώς ε, θα πρέπει να πλένουμε τα πιάτα. Ε, και έτσι δεν έγινε δεκτή η πρόταση της Επιτροπής να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής στα πλαστικά γάντια για την κουζίνα και δεν θα υπάρξει νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα προϊόντα αυτά. Επίσης δεν θα υπάρξει νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα προϊόντα που πολλούνται, που παράγονται στα σπίτια, τα τρόφιμα και πολλούνται στις χριστουγεννιάτικες ε, αγορές. Ε, δεν υπάρχει ανάγκη νομοθεσίας για τέτοιου είδους προϊόντα. Και δεδομένου ότι πολλές χώρες όπως και η δική μου ήδη έχουν ε, κάποιες προδιαγραφές αγοράς ε, για ορισμένα προϊόντα, δεν πιστεύω ότι ε, δεν πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ε, μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί εκατοντάδες τροπολογίες ε, για μια νομοθεσία η οποία στοχεύει στην ε, απλούστευση και στον εξυγχρονισμό της, του φυστάμενου συστήματος. Κυρία Στήλερ, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης ηγετές και τους συνεργάτες μου για την πρόταση κανονισμού όσον αφορά τι συσκευέ αερίου. Συσκευέ οι οποίε χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθημερινά για την παραγωγή του φαγητού ή για τη θέρμανση. Είναι πολύ σημαντικό να θεωρούμε όμως ότι οι συσκευέ αυτές είναι όντως ασφαλείς και ότι μπορούν ως ασφαλείς να πολλούνται παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα αυτή πρόταση καταδεικνύει ότι όταν συνεργαζόμαστε για να δημιουργούμε έναν κοινό κανονισμό για όλες αυτές τις γεφές αερίου, τότε μπορούμε να έχουμε την ύψιστη δυνατή ασφάλεια όλων αυτών των συσκευών που καλύπτουν 500 εκατομμύρια πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικές λοιπόν απαιτήσει όσον αφορά τη λειτουργία, όσον αφορά την ασφάλεια, οι οποίες πρέπει να είναι κοινέ σε όλα τα κράτη-μέλη. Αύριο θα ψηφίσουμε λοιπόν στην Ολομέλεια και θα καταλήξουμε σε ένα τελικό κείμενο μετά από πάρα πολύ καιρό που περάσαμε σε τριμερείς διαλόγους. Ελπίζω ότι θα καταφέρετε όλοι να εγκρίνετε το συμβαστικό αυτό κείμενο, το οποίο είναι, θεωρώ ότι είναι θετικό και καλύπτει όλες τις προτάσεις που γίνανε από όλε τις πλευρές. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να έχουμε ένα κανονισμό και μέχρι τον Ιανουάριο 2018 αυτό θα ισχύσει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύπτονται πάρα πολλά προϊόντα, θερμαντές, κουζίνες, και άλλες συσκευές. 476.000 άτομα χρησιμοποιούν τις ε, συσκευές αυτές και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι ε, έχουμε περίπου 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικό κύκλο εργασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα κατασκευής αυτών των συσκευών όταν διατίθενται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια τόσο των ανθρώπων όσο και των κατοικίδιων ζώων. Μιλώντας για υγεία και ασφάλεια θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε και το ζήτημα του μονοξιδίου του άνθρακα. Ξέρετε όταν τον φυσικό αέριο καίγεται, παράγει και μονοξίδιο του άνθρακα όταν αυτό έρχεται σε επαφή με το οξυγόνο που έχουμε στην ατμόσφαιρα. Το μονοξίδιο του άνθρακα είναι ιδιαίτερα δηλητηριώδες. Έχουν γίνει λοιπόν κάποιες συγκεκριμένε αναφορές στον κανονισμό αυτό και χαίρομαι πάρα πολύ που και στο τελικό κείμενο γίνεται ρητή αναφορά στον κίνδυνο δηλητηρίαση από μονοξίδιο του άνθρακα. Δυστυχώ όμω τα κράτη-μέλη δεν κάνουν ακόμα αρκετά πράγματα γι' αυτό και από ό,τι φαίνεται οι περισσότεροι δεν λαμβάνουν υπόψη του το πρόβλημα αυτό. 200 άτομα το χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο χάνουν ε, τη ζωή τους εξαιτία τη δηλητηρίαση από μονοξιδίου του άνθρακα. Θα μπορούσαμε να αποφύγουμε όλους αυτούς τους θανάτους. Υπάρχουν ε, πολλά παιδιά στον Ηνωμένο Βασίλειο τα οποία χάσαν τη ζωή τους, συγκεκριμένα περιπτώσεις το 2006 και επίσης είχαμε τέτοια φαινόμενα και σε ένα ξενοδοχείο στην Κέρκυρα, ακριβώ επειδή εκεί χρησιμοποιείται μία σόμπα η οποία δεν τηρούσε τα πρότυπα ασφάλειας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε πλέον ένα κανονισμό ο οποίος ευθυγραμμίζει τις διασφαλίσεις ασφάλειας αυτών των συσκευών παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το μονοξίδιο του άνθρακα σκοτώνει πολύ περισσότερους ανθρώπους ε, ετησίως από ότι το AIDS ή ο καρκίνος του δέρματος. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ευθυγραμμίσουμε το επίπεδο ασφάλειας των ξενοδοχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δυστυχώς αυτή τη στιγμή παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλη απόκληση. Σαφώς οι καταναλωτές θα πρέπει να προστατεύονται από πουδήποτε και αν μένουν, οπουδήποτε και αν πηγαίνουν διακοπές καθότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ε, προτάσεις όσον αφορά τα ξενοδοχεία, θα θέλαμε να υποστηρίξουμε τη σύσταση του Συμβουλίου του 1996 όσον αφορά τα και ασφαλεία στα ξενοδοχεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω όσον αφορά συσκευέ που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Εφόσον δεν υπάρχει λοιπόν κανένα αρμόδιο σχετικό κανονισμό, θα θέλαμε να έχουμε ένα κοινό σύστημα ανιχνευτών για το μονοξυδίου του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώ δεν έχουμε καν κάποιο παρατηρητήριο το οποίο να μπορεί να συλλέγει όλα αυτά τα δεδομένα για τι εκκλήσει, για τι εκροέ μονοξιδίου του άνθρακα από διάφορε συσκευέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμφωνήσετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα του φυσικού αερίου, ο κίνδυνος του μονοξιδίου του άνθρακα και θα πρέπει και για τα δύο αυτά ζητήματα να έχουμε κοινά πρότυπα, κοινέ προδιαγραφές παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Λόπες Ιστούριτς Βάιτ έχει τώρα το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ συνάδελφοι σε αυτό το καταπληκτικό ακροατήριο. 17.500 εγκαταστάσεις ε, με σειρματόσχηνα υπάρχουν στις Άλπεις και αλλού. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει δεσπόζουσα θέση στις μεταφορές με σειρματόσχηνο. Το 60% της παγκόσμιας αγοράς κατέχει. Η βιομηχανία του σκι είναι ο κλάδος ο βασικός, αλλά και αλλού. Μιλούμε για 4.000 θέσεις απασχόλησης από τις επιχειρήσεις που βάζουν αυτές τις εγκαταστάσεις με σειρματόσχηνα και έχουμε πάρα πολλούς χρήστες. Είναι σημαντικό να έχουμε προστασία του καταναλωτή και πλήρη εναρμόνιση των τεχνικών ε, προδιαγραφών με κανόνες αφής λεπτομερής που θα εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σήμα που θα είναι ποιότητας που θα πάει του ευρωπαϊκού προϊόν σε μια σφαίρα ανώτερη και καλύτερη. Όλα αυτά εντάσσονται στην ε, ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και την προστασία του καταναλωτή. Από το 1951 οπότε δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα. Η οικονομική ολοκλήρωση ήταν ο κινητήριος μοχλός για την ανάπτυξη των κοινωνιών μας. Εάν έχουμε εσωτερική αγορά έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη και ανάπτυξη των εταιριών μας πρέπει να τονίσουμε τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απόσταση που οφείλουμε να διανύσουμε για να δημιουργήσουμε πλούτο και ε, ανάπτυξη για τις επιχειρήσεις μας. Με αυτές τις τρεις εκθέσεις προχωρούμε σε μια αγορά ακόμα πιο ολοκληρωμένη, φιλική προς τους καταναλωτές και προς τις επιχειρήσεις. Η αγορά των εγκαταστάσεων με σειρματόσχηνα χαρακτηρίζεται από υψηλή εξειδίκευση και γι' αυτό η έκθεση αυτή έχει πάρα πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Η οδηγία του 2000 αντικαθίσταται με κανονισμό σήμερα και Αύριο θα καταργήσουμε τις αποκλίσεις μεταξύ κρατών μελών. Μπορούμε να έχουμε πλήρη εναρμόνιση και μπορούμε όλοι να τηρήσουμε την γενική πολιτική δέσμευση ε, που σημαίνει ότι εργαζόμαστε για καλύτερη νομική πλαισίωση και απλούστευση των νομικών διαδικασιών. Έτσι ε, εγκαταστάσεις ασφαλείας και συστατικά ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις με να θα είναι υποχρεωτικές, θα εγγυόμαστε αυτά τα προϊόντα και θα εφαρμόζεται με ομοιόμορφο τρόπο σε όλη την Ένωση η πλήρη εναρμόνιση. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να επιβάλλουν πιο αυστηρές προϋποθέσεις ή νέες και διαφορετικές προϋποθέσεις με, στην εθνική νομοθεσία και έτσι η βιομηχανία έχει την εγγύηση ότι το εμπόρευμά της στηρεί τις προϋποθέσεις και μπορεί να απολυθεί παντού και αποφεύγονται τα απαραίτητα ε, κόστη για την ενσωμάτωση μιας οδηγίας, αφού τώρα θα έχουμε κανονισμό. Και μιλούμε για την χωροταξία και για την προστασία του περιβάλλοντος και για τις χρήσεις γης. Όλα αυτά θα ωφεληθούν από τον κανονισμό. Ο νέος κανονισμός έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής και απαριθμεί τις εξαιρέσεις ξεκάθαρα και δίνονται διευκρινήσεις ως προς τις εγκαταστάσεις με σειρματόσχηνα για τη μεταφορά ατόμων και για τις δραστηριότητες αναψυχής. Αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής οι δραστηριότητες ε, αναψυχής σε πάρκα ε, με ατραξιόν και σε παντηγύρια εκεί υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις και πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει σύστημα αξιολόγησης για όλα τα ανταλλακτικά και κάνουμε το πάνω για να μην υπάρχει στρέβλωση της αγοράς και διαφορετική μεταχείριση. Και όλα αυτά τα οποία προβλέπονται ε, επεκτείνεται η προστασία και στα υποσυστήματα ασφαλείας. Ευχαριστώ να δώσω το λόγο στην, ε, στον, ε, στην Επίτροπο Μπιενκόφσκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, εξότιμα μέλη. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και να συγχαρώ τους εισηγητές, την κυρία Φόρντ, τον κύριο Στήλερ και την κυρία Λόπεθ Λόπαθη Βάιτ για την σκληρή τους εργασία σε αυτούς τους τρεις πυλώνες που οδήγησαν ε, σε, μια, σε, σημαντικά, σε θετικά αποτελέσματα. Ε, ε, και πραγματικά θα υπάρξουν αποτελέσματα. Είναι σημαντικό βήμα στην εξασφάλιση απλούστασης του νομικού πλαισίου. Τρεις κανονισμοί καλύπτουν ένα σημαντικό τμήμα, κομμάτι των προϊόντων τα οποία δικαινούνται στην εσωτερική αγορά και αφορούν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούν εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών σε καθημερινή βάση. Είναι σημαντικό μια, ένας ενιαίος ε, κανονισμός ε, της εσωτερικής αγοράς εξασφαλίζει την ε, ασφάλεια των προϊόντων ειδικά όσον αφορά τον προστατευτικό εξοπλισμό για τους εργαζόμενους. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε οι εταιρείε οι οποίες παράγουν αυτά τα προϊόντα μπορούν να βασιστούν σε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο πληρεί τις ανάγκες τους και τους επιτρέπει να είναι ανταγωνιστικές. Ένα νομικό πλαίσιο το οποίο είναι ξεκάθαρο και δεν επιβάλλει υπερβολικό άχθος, ε, υπερβολικά εμπόδια. Ε, Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση, πρόκειται για οδηγίες οι οποίες θα μετατραπούν σε κανονισμούς οι οποίοι θα είναι άμεσα εφαρμοστές σε όλες τις χώρες μέλη και αυτό θα διευκολύνει πάρα πολύ των, ε, της επιχείρησης. Γιατί αντί να υπάρχουν 28 διαφορετικά συστήματα μεταφοράς, οι εταιρείε θα μπορούν να αναφέρονται σε ένα μόνο ενιαίο κείμενο το οποίο θα διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι προσεγγίσουμε περισσότερο την ε, ολοκλήρωση του νέου κανονιστικού πλαισίου το οποίο θα προσδώσει μεγαλύτερη συνοχή στην ε, εσωτερική αγορά και θα είναι πιο εύκολα εφαρμόσιμο. Τώρα υπάρχει ένα πολύ ξεκάθαρο, μια ξεκάθαρη ε, δέσμη ε, δεσμεύσεων για τους ε, κατασκευαστές. Η διαδικασία ίχνηλασιμότητας θα μας βοηθάει να εντοπίζουμε τα προϊόντα σε, όλη την, σε όλο το μήκος της αλυσίδας. Επίσης οι υποπτικές αρχές θα μπορούν να καταπολεμήσουν πιο αποτελεσματικά μη ασφαλή προϊόντα που δεν συμμορφώνουν με τι προδιαγραφέ τη εσωτερική αγορά και αυτό θα είναι ει όλων των επιχειρήσεων, οι οποίε θα πρέπει να συμμορφώνονται με του εφαρμοστέου κανόνε. Και έτσι θα μειωθεί, θα συρρικνωθεί ο θέμητο ανταγωνισμό. Τα ωφέλη ε, αυτού του κανονισμού ε, ισχύουν ε, και για τους κατασκευαστές και για τους καταναλωτές. Και θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για το θεσμικό θέμα. Ε, γίνονται διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο ε, της διοργανική συμφωνίας και έχει επικυρωθεί ότι οι επιτροπολογίες δεν μπορούν να εξωθούν με τις ε, ομάδες εμπειρογνωμόνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με το ρόλο των επιτροπών. Κυρίες και κύριοι, έγκριση αυτών των προτάσεων θα έχει μια θετική επίπτωση στην επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη έτσι θεωρώντας ότι έχει επιτευχθεί μια συμφωνία από τους νομοθέτες και με τον τρόπο αυτό υπάρχει μια σημαντική προσθέμενη αξία για τους επιχειρηματίες αλλά και για τις δημόσιες διοικήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, χαιρετίζει αυτό το πακέτο των κανονισμών. Η κυρία Αζέα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ω εισηγήτρια γνωμοδότηση τη Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων, για αυτές τις τρει προτάσεις ε, κανονισμού και ιδίω για τα μέσα ατομική προστασία, πρέπει να σα πω ότι η δική μου γνωμοδότηση ομόφωνα εγκρίθηκε από την Επιτροπή Απασχόληση. Στείλαμε πάρα πολλές ενδείξεις προς την καθήλυνα αρμόδια επιτροπή γιατί θεωρούμε ότι το ζήτημα της ασφάλειας των εργαζομένων είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό. Είπαμε επίσης στη γνωμοδότησή μας ότι θα πρέπει να δοθούν τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, ανακλάδο και ότι θα πρέπει να ισχύουν κοινοί, κοινοί κανόνες, δηλαδή κοινή γλωσσική διατύπωση, κοινή ενημέρωση και πληροφόρηση κατανοητή για όσους χρησιμοποιούν τα μέσα τομικής προστασίας. Μας λυπεί όμως ότι η δική μας συμμετοχή της Επιτροπής Απασχόλησης δηλαδή δεν ήταν πάρα πολύ σημαντική και οι σημαντικότερες δικές μας ενδείξεις ως προς την ενημέρωση και την πληροφόρηση για τη χρησιμοποίηση των μέσων, μέσων αυτών ατομικής προστασίας τελικά δεν ελήφθη σοβαρά υπόψη από την καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Νομίζω ότι ε, είναι πολύ σημαντικό τελικά να δούμε ποια θα είναι η τελική μορφή που θα πάρει η έκθεση αυτή προτού δώσουμε εμείς την τελική μας έγκριση. Ο κύριος Σαγημό έχει το λόγο. Ξότιμοι συνάδελφοι, μελός ε, επικεφαλής αντιπραγματεύσεων εκ μέρου του ΕΛΚ για την πρόταση ενός κανονισμού για τον ε, προσωπικό εξοπλισμό. Η ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά χαρακτηρίζεται από υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και θα έλεγα πουθενά οι καταναλωτές δεν προστατεύονται τόσο αποτελεσματικά όσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα ο κανονισμός αυτός ε, αφορά πολύ υψηλές προδιαγραφές σε κάσκες κλπ. Δεν πρόκειται για, ε, ε, για πλαστικά γάντια. Και αν αγοράζω για την ε, κόρη μου μια κάσκα για το ποδήλατο, ε, ένας εργαζόμενος αγοράζει ένα προστατευτικό εξοπλισμό για την εργασία του ε, θα πρέπει να μπορεί να βασιστεί σε προϊόντα υψηλής ποιότητας. Για μας το ΕΛΚ ήταν σημαντικό επίσης να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να εφαρμόσουν άμεσα αυτές τις νέες διαδικασίες και χωρίς μεγάλο γραφειοκρατικό άχθος γιατί τι χρησιμεύουν και οι καλύτερες διατάξεις αν στη συνέχεια δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Και στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζω κυρίως τη συμφωνία για μια απλούστευση διαδικασίας ε, πιστοποίησης. Εάν ένας ε, κατασκευαστής δεν αλλάξει το προϊόν αλλά το προϊόν αυτό ε, ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να πληρώσει και πάλι για το, να καταβάλει το αντίτιμο του πιστοποιητικού άλλη μια φορά ε, θα πρέπει να καταργήσουμε τις ε, υπερβολικές γραφειοκρατικές αξιώσεις. Και υπό το πνεύμα αυτό θεωρώ την έκθεση θετική. Ε, κύριε Βέσφαλ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. η ατομική προστασία δεν είναι κάτι με το οποίο εμείς οι βουλευτές ε, θα καρποθούμε σημαντική αναγνώριση εκ μέρους της κοινή γνώμης. Ε, παρόλα αυτά είναι ένα σημαντικότατο θέμα γιατί ο προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες, ε, τα κράνη κλπ. ή για τους, για τους υπόλοιπους κλάδους ε, ε, ε, δεν πρόκειται μόνο για προστατευτικό εξοπλισμό για επαγγελματίε, αλλά και για ιδιωτική χρήση. Πρόκειται και για τα γάντια που χρησιμοποιούμε στο φούρνο και αυτά θα πρέπει να είναι ασφαλή. Και θεωρώ ότι αυτό το πετύχαμε στις διαπραγματεύσεις τόσο με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί πάντοτε είχαμε συνείδηση του κινδύνου να είμαστε υπερβολικά γραφειοκρατικοί. Γι' αυτό εξαιρέσαμε για παράδειγμα την αθλητική ενδυμασία ή τα πλαστικά γάντια για το πλήσιμο των πιάτων. Ε, θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα είναι καλό ε, και τόσο οι όσο και οι κατασκευαστές αλλά και οι υποπτικές αρχές της αγοράς ε, με τον κανονισμό αυτό έχουν ε, ένα, ε, μια πολύ καλή βάση. Ο κύριος Ντάλτον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλωσορίζω την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις εγκαταστάσεις με σειρματόσχηνα. Θα απλουστευτεί η γραφειοκρατία. Τα κράτη-μέλη θα μπορούν να ελέγξουν καλύτερα το κατά πόσο πληρούνται οι συνθήκες ασφαλείας και ούτω καθεξής. Χαίρομαι που αποκλείστηκαν τα ιστορικά σύρματόσχηνα από το πεδίο εφαρμογής. Έχουμε τον Βρετανικό σιδηρόδρομο που αρχικά ήταν ένας τρόπος να βοηθήσει τους ντόπιου να, ανέβουν, ε, να ανεβάσουν εμπορεύματα ή να ανέβουν οι ίδιοι σε ένα ύψος που θα ήταν πάνω από 200 σκαλοπάτια. Το να πρέπει οι ιστορικοί σιδηροδρομοί να συμμορφωθούν στους σύγχρονους κανονισμούς είναι κάτι το πολύ δυστυχές γιατί έχουν ιστορική αξία. Χαίρομαι διότι σε αυτή την περίπτωση δεν υιοθετήσαμε την προσέγγιση ένα μέγεθος να ταιριάζει σε όλους και τελικά οι μελλοντικέ γενιές θα μπορέσουν να απολαύσουν αυτό το σιδηρόδρομο στο Κλίφορντ. Ευχαριστώ κυρία Σαρανσόβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Αυτές οι, αυτοί οι τρει αυτοί οι τρεις φάκελοι δεν είναι και τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα, ειδικά αυτή την ώρα που είναι τόσο αργά. Όμως, χάρη στη δουλειά τη δική μας, ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα είναι λίγο πιο ασφαλής μετά την υπερψήφιση αύριο. Μπορεί να ξέρει ο Ευρωπαίος πολίτης ότι όταν πάει στη δουλειά του, όταν κάνει ένα ζεστό ντους, όταν παίρνει τον αναβατήρα για να κάνει σκι, ότι θα ξέρει ότι οι υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας ισχύουν και εφαρμόζονται. Χαίρομαι γιατί επικράτησε η κοινή λογική σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και έτσι οι ιστορικοί σιδηρόδρομοι με σειρματόσχηνα όπως αυτό στην Πράγα αποκλείονται από τον κανονισμό. Για εμένα αυτή η φάκελη είναι ένα καλό παράδειγμα του τι μπορεί να κάνει η ευρωπαϊκή εναρμόνιση. Αν δεν υπάρχει επαρκώς τεκμεριωμένος λόγος που να δικαιολογεί διαφορετικά στάνταρ, διαφορετικά πρότυπα από το μία χώρα μέλος στην άλλη, τότε ε, η εναρμόνιση ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και κάνει τη ζωή μας ευκολότερη. Κυρία Επίτροπε, θα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να ασκεί νομοθετική εξουσία για να εναρμονίσει εκεί που ε, είναι αυτολογικό και όπου τα ωφέλη είναι σαφέστατα. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για την εύρεθμη λειτουργία της εσωτερικής ενίας αγοράς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. κύριος Μαστάλκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε αγαπητοί συνάδελφοι. Κρίμα που κάνουμε τη συζήτηση αυτή τόσο αργά στην ημέρα και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά τόσο αργά, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να αντικαταστήσει τον προηγούμενο κανονισμό του 1999 και να έχει πλέον ομοιόμορφη εφαρμογή με τους νέους αυτούς κανονισμούς σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε επίσης ότι ε, ιδίως όσον αφορά τα μέσα ατομικής προστασίας μιλάμε για μια αγορά που αντιστοιχεί σε δισεκατομμύρια ευρώ σε τήσια βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης ένα τομέα ο οποίο γνωρίζει υψηλό επίπεδο καινοτομία. Χρησιμοποιούνται νέα ευφυή υλικά στον τομέα αυτό. Θεωρώ ότι οι προτάσεις που γίνονται εν γέννη είναι θετικέ, υπάρχουν όμω και κάποιε προβληματικές, όπως ε, για παράδειγμα η συμπερίληψη μέσω τομικής προστασίας για τη θέρμανση, το νερό. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα ισχύουν διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικοί ώρα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τις δηλώσεις συμμόρφωσης ή τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να πετύχουμε την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των καταναλωτών και την προστασία των κατασκευαστών και πώς μπορούμε βέβαια να αποφύγουμε τα εργατικά ατυχήματα. Πιστεύω πάντως ότι ο κανονισμός αυτός εν γέννη θα είναι πολύ θετικός για την ασφάλεια των πολιτών μας. Η κυρία Πάρκερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η εναρμόνιση, στην Ευρω... εναρμόνιση και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έννοιες οι οποίες πηγαίνουν μαζί. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα τρει προτάσει οι οποίε συμβάλλουν στην αύξηση τη εναρμόνιση στα κράτη-μέλη. Η προσέγγιση όμω τη κοινή λύση ε, για όλα δεν είναι θετική και αυτό το βλέπουμε και εδώ πέρα. Η κυβέρνηση του Μένου Βασιλείου έχει εκφράσει ανησυχίες όσον αφορά τον κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας και έχει ήδη πει ότι τίθεται κατά της πρότασης αυτής κανονισμού. Βέβαια το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγκαστεί να εφαρμόσει αυτόν τον κανονισμό. Συμφωνούμε βέβαια ότι προκειμένου να έχουμε μια αποτελεσματική αναγνώριση ανάμεσα στα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουμε και κοινού κανόνες, αλλά δεν ξέρω αν η ευθυγράμμιση είναι η καλύτερη λύση. Εγώ δεν είμαι ο κύριος Μπουζό έχει το λόγο. Κύρια Πρόεδρε, αξιότιμε κυρίες και αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την ε, κυρία Στέιλερ ιδιαίτερος, αλλά να συγχαρώ και τους τρεις ε, εισηγητές, γιατί πραγματικά το έργο τους ήταν εξαιρετικό ο νέος ε, κανονισμός για τις συσκευές ε, αρίου ε, μπορεί να είναι υποδειγματικό όσον αφορά την εναρμόνιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και εγκαιάται την ασφάλεια των συσκευών αυτό ε, αυτό ε, και εξασφαλίζει επίσης και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Πρόκειται για προδιαγραφές υψηλού επίπεδου που αφορούν την ασφάλεια των καταναλωτών και με τον τρόπο αυτό ε, μειώνονται τα, οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και επίσης έχουμε μια πιο ορθολογική χρήση της ενέργειας. Ε, αυτό αφορά τόσο μικρές φορητές οικιακές συσκευές αλλά και ε, λέβητες ε, πολυκατοικιών. Και αυξάνεται συνεχώς ο όγκος πωλήσεων συσκευών αερίου. Η συγκήτρια κυρία Στάιλερ αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα σε σχέση πάντα με την ασφάλεια των ε, καταναλωτών και Επίσης, ε, το πώς θα πρέπει να αποφευθούν οι δηλητηριάσεις από μονοξίδιο του άνθρακα, αλλά και από άλλες ε, τοξικές ουσίες. Οι δηλητηριάσεις από το μονοξίδιο του άνθρακα είναι σημαντικό αίτιο θανάτου κατά την χρήση συσκευών αερίου. Και τώρα ελπίζουμε θα εξαλειφθούν αυτοί οι κίνδυνοι. Κυρία Κόμη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, καλησπέρα σας. Η πραγματοποίηση της ιστορικής αγοράς είναι σαφώς σημαντική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταβάλουμε και πάρα πολλές προσπάθειες. Γι' αυτό συμφωνώ, αυτό κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η ευθυγράμμιση των εθνικών κανονισμών σε διάφορους τομείς αποτελεί σημαντικό βήμα της όλης αυτής διαδικασίας για την απλούστευση της κοινοτικής νομοθεσίας, η οποία όμως θα πρέπει να οδηγεί και σε καλύτερη προστασία των πολιτών, να βελτιωθεί δηλαδή η ζωή των πολιτών μας μέσω των κανονισμών αυτών και αυτό θα πρέπει να είναι στόχος μας. Όσο αφορά τη στρατηγική για την εσωτερική αγορά της υπηρεσίες και τα αγαθά για την οποία υπήρξα εισηγήτρια, θεωρώ ότι θα πρέπει να προωθήσουμε την προσέγγιση αυτή ουσιαστικά, να μην έχουμε πλέον συγκεκριμένα εμπόδια όσον αφορά την εναρμόνιση διαφόρων συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για οικονομική ένωση πάρα πολύ συχνά, αλλά δεν νομίζω ότι βλέπουμε παντού τελικά αυτή την οικονομική ένωση σε όλες τις πτυχές της. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να προχωρούμε με ευθυγράμμιση και να καταρρύπτουμε όλα τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν όσον αφορά τη χρησιμοποίηση κοινών προτύπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε με τι τρει προτάσει κανονισμού. Καλύτερη ευθυγράμμιση, περνάμε πλέον από οδηγίε σε κανονισμού. Αυτό είναι σίγουρα ένα βήμα πρόοδου και το να γνωρίζουμε αυτό σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει και εσεί να χρησιμοποιείτε όλο και περισσότερο τη μέθοδο αυτή. Θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό να έχουμε όλο και πιο συχνά κανονισμούς που θα εγκρίνονται με το συντομότερο δυνατό τρόπο. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δυναμώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και στι τρει αυτέ εκθέσει αναφερόμαστε σε διαφορετικού κλάδου, σε διαφορετικού τομεί, οι οποίοι όμω είναι πάρα πολύ σημαντικοί και για την οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι βελτιώνοντας τους κανόνες θα έχουμε θετικές επιπτώσεις και για την οικονομική ανάπτυξη αλλά και για την απασχόληση, ζητήματα που μας απασχολούν σε καθημερινή βάση. Ο κύριος Ρούμπιχ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω ότι το θέμα εδώ είναι μέσω της εναρμόνισης να πετύχουμε και οικονομικά εφέλη, ιδιαίτερως για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ρυθμίζοντα και τι δυνατότητε πρόσβασης στην αγορά. Επίσης είναι ξεκάθαρο ότι ο κανονισμός ε, για τις ε, εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις, παίζει σημαντικό ρόλο στον τουρισμό. και για παράδειγμα τα τελεφερίκ μελλοντικά δεν θα επιβαρύνουν καθόλου την ε, ατμόσφαιρα με και, θα εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Ε, Αποδεικνύεται έτσι ότι η Ευρώπη μπορεί να αξιοποιήσει τα ωφέλη της εσωτερικής ε, αγοράς δημιουργώντας και νέες θέσεις απασχόλησης. Για αυτό το νέο ήθος ε, πολιτικής ε, ασφαλείας ανοίγει το δρόμο και στους κατασκευαστές συμβάλλοντας καθοριστικά και στα επίπεδα ασφαλείας. Η ε, κατασκευάστερες εταιρείες με τον τρόπο αυτό έχουν ένα ε, αυξήσει το κύκλο εργασιών και τα μέσα, αυτής, τα μέσα αυτά μεταφοράς θεωρούνται πλέον πολύ σημαντικά καθώς, ε, διότι έχουν και έναν πολύ υψηλό βαθμό βιωσιμότητας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας για το θέμα αυτό. Πράγματι δεν είναι ένα θέμα που καταλαμβάνει την πρώτη σελίδα στις εφημερίδες, αλλά είναι σημαντικό για τους καταναλωτές. Και χαίρομαι γιατί έχουμε βουλευτές που δίνουν ενέργεια, δίνουν χρόνο και εμπειρογνωμοσύνη για αυτό το θέμα. Η δουλειά τους θα σώσει ζωές χάρη στα πρότυπα τα εναρμονισμένα. Χάρη στο ότι όλα θα γίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Και στα μέσα ατομικής προστασίας και στις συσκευές αερίου και στις εγκαταστάσεις με σειρματόσχηνα. Στη χώρα μου Έχουμε ένα μικρό νησάκι που εξαρτάται από ένα σειρματόσχηνο μέσα από το οποίο συνδέεται με την ενδοχώρα. Ως προς τις συσκευές αερίου. Έχουμε 30 εκατομμύρια ε, κουζίνες, φούρνους, σόμπες, μπόιλερ στην Ευρώπη και όλα αυτά μπορεί να δώσουν λαβή για ατυχήματα με την έκκληση μονοξυδίου του άνθρακα. Και είχαμε μια πολύ σημαντική εκστρατεία συνειδητοποίησης και ε, ενημέρωσης για το μονοξίδιο του άνθρακα. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και μας βοηθούν να ε, πάμε στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Για τα μέσα ατομικής προστασίας πρέπει να ακούσουμε τη βίκη Ford που μας έδειξε τι μπορεί να γίνει με τα κατώτερης ποιότητας προϊόντα όταν αυτά μπαίνουν στην αγορά. Πρέπει να έχουμε κοινά πρότυπα και να διασφαλίσουμε ότι εφαρμόζονται. Αυτό θα ενθαρρύνει και τους παραγωγούς να συμμορφωθούν με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και θα καθησυχάσει τους καταναλωτές ότι έχουν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα και στα μέσα ατομικής προστασίας και στις συσκευές που αγοράζουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος ε, Τσίριο παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι σήμερα κάνουμε μία συζήτηση η οποία είναι τελικά πολύ σημαντική και έχει να κάνει με πάρα πολλά υλικά, με πάρα πολλές συσκευές, όχι μόνο αυτές που παριθμούνται στα έγγραφα που έχουμε ενώπιον μας. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια σημαντικότατη εναρμόνιση που γίνεται σε πάρα πολλούς τομείς. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, θα ήταν σκόπιμο ήδη να αρχίσουμε να ρωματιζόμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με κοινού κανόνες, όπου όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, θα χαίρουν ισότιμων ε, ποιοτικών προϊόντων. Σήμερα, πιο συγκεκριμένα, ψηφίζοντας και συζητώντας σε αυτή την ολομέλεια την εναρμόνιση των προτύπων όσον αφορά τις εγκαταστάσεις με σειρματόσχηνα και να φέρουμε εδώ πέρα κυρίως τις ορεινές περιοχές που χρησιμοποιούν τελεφερίκ θεωρώ πραγματικά ότι ενεργούμε υπέρ όλων αυτών των κέντρων, χιονοδρομικών κέντρων κτλ. Οποιουσδήποτε γνωρίζει λίγο για τα κέντρα αυτά θα γνωρίζει τελικά ότι πρόκειται συνήθως για χινοδρομικά κέντρα τα οποία βρίσκονται πολύ μακριά το ένα από το άλλο αλλά πέρα από τη γεωγραφική απόκληση υπάρχει και μια τεχνική απόκληση. Οι κέντρα της Ιταλίας και της Γαλλίας δεν έχουν τα ίδια πρότυπα. Θεωρώ λοιπόν ότι σήμερα κάνουμε ένα σημαντικότατο βήμα πρόοδου. Είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε όλο και περισσότερο τέτοιες εκθέσεις που συμβάλλουν στην αρμόνιση πολλών κλάδων και άλλωστε τους κλάδους θα πρέπει να αρμονίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μόνο έτσι πετυχαίνουμε και οικονομική ανάπτυξη. Ο κύριος Ποσπισίλ έχει το λόγο, είναι το τελευταίο ομιλητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τους προλύσαντες, λέγοντας ότι εντάξει, έχουμε καλύψει τα περισσότερα πράγματα όσον αφορά τις τρεις αυτές εκθέσεις. Να πω πάντως και εγώ ότι θεωρώ ότι σημειώνουμε ένα σημαντικό το βήμα πρόοδου και απευθυνόμενο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πω ότι αυτό το οποίο εκ πρώτης όψεως πρέπει να φαίνεται ως μια καθαρή τυπικότητα, το ότι περνάμε από μια οδηγία σε ένα κανονισμό, στην πράξη δεν αποτελεί απλώς τυπικότητα. Εγώ ήμουν υπεύθυνο για τη δικασία αυτή στην Τσεχία και γνωρίζω πολύ συχνά ότι οι οδηγίες μπορεί να οδηγήσουν σε 6, 8, 10 διαφορετικούς εφαρμοστικούς νόμους. Επομένως, αν πραγματικά θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων, ε, τότε είναι πολύ θετικό να πετυχαίνουμε τέτοιες συμφωνίες για κανονισμούς, οι οποίοι ομοιόμορφα εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλα τα κράτη-μέλη. Σημαντικότατο λοιπόν το βήμα αυτό προόδου Προς το συγκεκριμένο περιεχόμενο των κανονισμών αυτών θεωρώ ότι και το περιεχόμενό τους και οι λεπτομέρειές τους είναι πολύ καλύτερες σε σχέση με τα στοιχεία τα οποία είχαμε στις αντίστοιχες οδηγίες. Νομίζω ότι πάρα πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες θα αποφεληθούν από τους ομοιόμορφους αυτούς κανόνες, αυξάνεται το επίπεδο ασφάλειας, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στην εκπόνηση των εκθέσεων αυτών και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό το ότι έχουμε τις τρεις αυτές προτάσεις. Περνάμε τώρα σε διαδικασία Catch the Eye. Το λόγο έχει ο κύριος Μαριάς. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συζητούμε ένα πάρα πολύ σοβαρά θέμα το οποίο έχει σχέση και με την ασφάλεια των καταναλωτών αλλά και την ασφάλεια των ίδιων των εργαζομένων. Και είναι προφανές ότι η οικονομική παγκοσμιοποίηση και η απελευθέρωση του εμπορίου είχαν σαν αποτέλεσμα την μεταφορά της παραγωγής στις αναπτυσσόμενες χώρες εκεί όπου προκειμένου να μειωθεί το κόστος και να έχουν οι επιχειρήσεις μεγαλύτερο κέρδος είχαμε ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι προδιαγραφές ασφαλείας. αποτέλεσμα ήταν λοιπόν να έχουμε πάρα πολλά ε, εμπορεύματα και συσκευές στην ευρώπη οι οποίες να είναι επικίνδυνες ιδίως συσκευές αερίου οι οποίες ήταν εισαγόμενες από την κίνα και είχαμε πάρα πολλά δυστυχήματα ιδίως λόγω της έκρησης του μονοξιδίου του άνθρακα μάλιστα σε χώρες με ενεργειακή φτώχεια όπως η ελλάδα η οποία έχει χτυπηθεί από το μνημόνιο δυστυχώς είχαμε και τέτοια συμπτώματα. είναι σημαντικό που λαμβάνονται αυτά τα μέτρα. ευχαριστώ. Now, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ για όλα σας τα σχόλια, για αυτή τη δέσμη, για αυτό το πακέτο. Για πρώτη φορά στην ε, βραχία με εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή άκουσα τόσο πολλές ε, ομόφωνα θετικές ε, γνώμες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους εγητές που συνεργάστηκαν τόσο στενά και εξασφάλισαν συνοχή στα τρία αυτά κείμενα καθώς και με το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Θα ήθελα να υπογραμμίσω εδώ τρία βασικά σημεία. Με αυτούς τους τρεις ε, κανονισμούς θα έχουμε έναν πιο απλουστευμένο και εξυγχρονισμένο νομικό πλαίσιο θα διευκολυνθεί ο βίος των ε, επιχειρηματιών και θα υπάρξουν πιο ασφαλή προϊόντα, κάτι βασικό για τους ε, πολίτες. Και πάλι λοιπόν θα ήθελα να σας παρακαλέσω να στηρίξετε το, τη δέσμη αυτών των τριών κανονισμών. Και τώρα θα έρθουμε στους ηγητές. Η κυρία Φόρντ έχει πρώτο λόγο. Thank Μία ενιαία αγορά θα πρέπει να διευκολύνει το βίο των καταναλωτών. Και ορισμένε φορέ ε, δεν χρειαζόμαστε μία ενιαία προσέγγιση, αλλά ορισμένε φορέ χρειαζόμαστε μία ενιαία κοινή λύση. Ε, οι πολιτε θα πρέπει να είναι ε, ασφαλεί έναντι του κινδύνου αξίδιου του άνθρακα. Ε, ούτως ώστε επίσης ε, να μην ε, πεθαίνουν από τραυματισμούς επειδή καταστρέφεται η καρέκλα στην οποία κάθονται, σπάει. Είναι σημαντικό να έχουμε έναν απλουστευμένο κανονισμό εδώ. Κάναμε, μια πολύ καλύτερη θέση και στη δική μου έκθεση εγώ κατέθεσα 146 τροπολογίες, 117 από αυτές ε, περιλήφθησαν ε, στον κανονισμό, ούτως ώστε να διευκολύνουμε ε, την ε, λειτουργία των ε, μικρότερων επιχειρήσεων, να μειώσουμε το γραφειοκρατικό άχθος και να μην αυξήσουμε το κόστος για τους καταναλωτές και τους κατασκευαστές. Ε, συνάδελφος αυτό ο ΚΙΠ είπε ότι δεν κατανοεί γιατί χρειαζόμαστε μια τέτοιου είδους νομοθεσία δεν κατέθεσε ούτε μία τροπολογία. Όταν το ζητούμενο είναι να εκπονηθεί η νομοθεσία, ε, εγώ θα προτιμούσα να συμμετάσχει κανείς ενεργά στο τραπέζι των ε, διαπραγματεύσεων. Ευχαριστούμε κυρία Στήλερ, έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές. Ακούσαμε όντως πολύ θετικά ενθαρρυντικά σχόλια από τους συναδέλφους, με συγκινεί ιδιαίτερα αυτό και πραγματικά συντοπεί κανείς ότι κάνουμε μια συγκεκριμένη δουλειά που πολλές φορές σώζει και δουλειές, ε, ζωές, με συγχωρείτε. Καταλαβαίνετε λοιπόν για ποιο λόγο καθόμαστε τόσο αργά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όσον αφορά την ενιαία αγορά, η Βίκη έχει απόλυτο δίκιο. Συνεργαζόμαστε, καταλήγουμε σε συμβαστικές λύσεις, αν ε, το UKIP είχε πάρει το πάνω χέρι σε αυτή τη διαδικασία, ότι η διαπραγμάτευση θα είχε γίνει, θα μας λέγανε απλώς να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα πρότεινε κανένα μία εμπρακτή λύση, ούτε θα προστάτευε τις ανθρώπινες ζωές. Πρέπει λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο, το λέω και αυτό, να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η προηγούμενη Ολλανδική Προεδρία πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν ξανά είχαν δηλαδή την Προεδρία στο παρελθόν, είχαν πει ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί κάποιες πολύ συγκεκριμένε διαδικασίες, πολύτιμες όμως, τις οποίες θα πρέπει να προασπίσουμε. Το ότι έχουμε καταλήξει αυτή τη στιγμή σε μια νέα αγορά με 500 εκατομμύρια καταναλωτές σε 28 κράτη-μέλη και μπορούμε αυτή τη στιγμή να λαμβάνουμε αποφάσεις υπέρ όλων αυτών των ανθρώπων, αποφασίζοντα κάτι θετικό για όλους αυτούς τους πολίτες, αν μη τι άλλο αυτό δεν έχει αξία, είναι ιδιαίτερα πολύτιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για τη συνεργασία σας, ευχαριστώ πάρα πολύ πολύ που θέλετε κι εσείς η εσωτερική αγορά να υπάρχει και να λειτουργεί υπέρ των πολιτών μας. Ο κύριος Λοπές Ιστούριτς Βουάιτ είναι ο τελευταίος ομιλητής μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους. Νομίζω ότι είναι κοινή η δουλειά συλλογική και χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με την κυρία Φόρτ και την κυρία Στήλερ. Μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσει, πάντοτε κάποιοι θέλουν να μην συμμετέχουν, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι δουλέψαμε οι περισσότεροι πολύ ικανοποιητικά και γίνεται ένα τεράστιο βήμα στην εσωτερική αγορά. Και γι' αυτό εγώ θέλησα να είμαι μέλο αυτή τη Επιτροπή. Είμαι νέο μέλο τη Επιτροπή και είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με την κυρία Φόρτ και την κυρία Στήλερ, από τι οποίε έμαθα πάρα πολλά. Να σα απαριθμίσω τέσσερα σημαντικά στοιχεία για την τελική έκθεση, ε, ε, την οποία είχα τη τιμή να συντάξω. Περισσότερο περισσότερη ενημέρωση και πληροφόρηση για τους καταναλωτές. Αναφορά στη διαδικτυακή τοποθεσία των ε, παραγωγών. Ε, ρυθμίσεις για το σύστημα πέδησης στις μεταφορές με σύρματόσχηνα. Και έτσι θα έχουμε πραγματικό ανταγωνισμό, νέα αιτιολογική σκέψη για τις κυρώσεις, και θέλω να αναφέρω εδώ τη σκιώδη εισηγήτρια κυρία Λούση Άντερσον που επέμεινε ιδιαιτέρως και έτσι έχει ενισχυθεί το σύστημα κοινώσεων του κανονισμού και τέλος ε, ε, μέρημνα για τις ιστορικές εγκαταστάσεις με αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον. Το ΕΛΚ είναι υπεύθυνο για αυτή την έκθεση και θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδης εισηγητές και αυτό μας επέτρεψε όλες τις τροπολογίες που εντάσσονται στο πεδίο αρμοδιότητας της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής να τις αξιολογήσουμε σωστά και μπορούμε να είμαστε περήφανοι ως μέλη της Επιτροπής ΙΜΚΟ. Ευχαριστώ σε όλους. Καλό βράδυ. Η Πρόεδρος. Και εγώ σας ευχαριστώ.